μια προφορική ερώτηση με θέμα τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Αρχικά την έχει υποβάλει η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπεάρτερ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε ενώπιον μας σήμερα ως μία από τις εισηγήτριες για την οδηγία κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Χαίρομαι που θα σας, ακούσαν, θα σας ακούσουμε. Εμείς έχουμε καλά ανθρώπινα στοιχεία για την αντιμετώπιση της εμπορίας των ανθρώπων. Η ε, οδηγία του 2011 αποτελεί μέτρο για την ε, προστασία των θυμάτων. Όμως η φύση του εγκλήματος ε, μας οδηγεί στο να μην έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Η Eurostat έκρινε ότι μεταξύ 2010 και 2012 είχαμε 30.000 θύματα σε 28 κράτη-μέλη, το 80% των οποίων ήταν γυναίκες. Βεβαίως αυτά τα στοιχεία δεν αναφέρονται στα θύματα, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, παρόλο που ελέγχονται και κρατούνται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως υπάρχει η διάσταση του φύλου σε αυτά τα εγκλήματα. Το 69% έτυχαν, ήταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ε, και το μεγαλύτερο μέρος ήταν οι γυναίκες. Άρα όσο σωστή και να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ε, επικαθίσουμε στις ε, δάφνες μας. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι αυτή η εργασία ε, δίνει πολλά κέρδη στους διακινητές. Γιατί λοιπόν δεχόμαστε το ότι οι εθνικές αρχές δεν αναλαμβάνουν άμεση δράση. Γιατί δεν διώκονται για το γεγονός ότι δεν σας έχουν δώσει τα σωστά αριθμητικά στοιχεία και δεν αντιμετωπίζουν την διακίνηση αυτή, ενώ άλλες χώρες ε, δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία και δεν αναγνωρίζουν αυτά τα εγκλήματα με σπουδή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ε, διώξουμε τους διακινητές και να υπερασπιστούμε τα θύματα πώς μπορούμε, πόσο πρέπει να περιμένουμε πλέον έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ε, πολλούνται σαν να ήταν ένα σακί πατάτες θα βρουν το δίκιο τους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στο θέμα, γιατί η διακίνηση ανθρώπων είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχησή μας, αλλά θα πρέπει να δούμε τα αίτια της κακοδαιμονίας και να διώξουμε τους διακινητές εάν μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στις χώρες υποδοχής και στις ε, χώρες ε, προέλευσης. Μετά το 2016 με αυτή τη στρατηγική θέλουμε να εξαλείψουμε τη διακέτη την εμπορία τους. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί σας για να καταπολεμήσουμε αυτό το ιταμό εμπόριο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία κατά της εμπορίας των ανθρώπων σε κάθε κράτος μέλος. Ελπίζουμε ότι η εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Η διακίνηση των ανθρώπων έχει σαν στόχο τους πιο ευάλωτους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε, για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα αυτό, ποια είναι η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Μιλάμε για, μιλήσαμε για την μετανάστευση και τους ε, πρόσφυγες, αλλά πραγματικά η διακίνηση των ανθρώπων είναι ένα ιταμό έγκλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ελπίζουμε, ε, κύριε Επίτροπε, τους επερχόμενους μήνες να αντιμετωπίσουμε αυτό το έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίζω τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την κυρία Μπεάρντερ που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία υποβολής της προφορικής ερώτησης. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, θερμά ε, για το σταθερό και έντονο ενδιαφέρον σας ε, να ασχοληθείτε με την εμπορία ανθρώπων και να τη βάζετε πάντα στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλούμε για εμπορία ανθρώπων, μιλούμε ουσιαστικά για αγοραπολισία ανθρώπων και των υπηρεσιών τους. Η εμπορία των ανθρώπων απαγορεύεται ρητά στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπιση ε, της ε, εμπορίας ε, γίνεται για να διορθωθεί αυτή η καταπάτηση. Επίσης, αποτελεί μια σοβαρή μορφή εργονομένου εγκλήματος, όπως προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αυτό το επονίδιστο και απεχθές έγκλημα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν τεράστια κέρδη για τους διακινητές από τέτοιες μορφές εκμετάλλευσης. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε περισσότερα θύματα των διακινητών, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τους διάβλους ε, των χρημάτων και στους νόμους και παράνομους τομείς και να σταματήσουμε να διακόψουμε αυτές τις ροές των χρημάτων. Η εμπορία των ανθρώπων αποτελεί πια ένα αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, αλλά και του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα φαινόμενο με σαφείς διασυνδέσεις ε, με πολλές πολιτικές ε, και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία της Eurostat ε, μας δείχνουν ότι για το 2010-2012 στις 28 χώρες μέλη έχουν καταγραφεί 30.146 θύματα της εμπορίας ανθρώπων. 80% των θυμάτων αυτών είναι γένους θηλυκού και 70% των διακινητών είναι άνδρες. 16% των δηλωμένων θυμάτων, των καταγεγραμμένων θυμάτων είναι παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Αυτά δείχνουν ότι η πιο εκτεταμένη και δεδομένη μορφή εκμετάλλευσης είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, 69%. Οι γυναίκες και τα κορίτσια δυστυχώς αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 95%. Πάνω από 100.000 ε, παιδιά έτυχαν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ε, κατάφορα μία έντονη διάσταση φύλου στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια διαρθρωτική μορφή βίας εις βάρος των γυναικών και εμποδίζει σοβαρά την ικανότητα των γυναικών να απολαύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους ε, επίσης όρις με τους άνδρες. Η διάσταση του φύλου διαδραματίζει ρόλο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της εμπορίας. Αυξάνει την ευπάθεια απέναντι στους διακινητές, ενισχύει την εκμετάλλευση και κρίνει η λιδία των μέτρων της συνδρομής και της βοήθειας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανο γιατί η Ευρωπαϊκή, Υπηρεσία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πολλά και ιδιαίτερα οι υπηρεσίε μου ασχολούνται με ιδιαίτερε φιλοδοξίε στον τομέα αυτό. Έχουμε πια ένα συνεκτικό νόμιμο ε, ένομο πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής που μας καθοδηγούν στις πολιτικές μας ε, για να πατάξουμε την εμπορία των ανθρώπων. Προσπαθούμε να κρυζώσουμε αυτό το φαινόμενο, όπως φαίνεται και στο πρόγραμμα για το 2012-2016. Η οδηγία για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων ε, έχει ως επίκεντρο τα θύματα και τα δικαιώματα. Επίσης, ε, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των παιδιών και στο θέμα της διάστασης του φύλου. Και η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας ε, εξέπνευσε στις 6 Απριλίου του 2013 χωρίς καθυστέρηση η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Ευρωπαϊκών Συνθήκων ξεκίνησε διαδικασίες ε, επιβολής κυρώσεων και με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι σήμερα 25 χώρες μέλη έχουν επίσημα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν μεταφέρει πλήρως την οδηγία αυτή στις εθνικές ένωμες τάξεις τους. Και μόνο δύο χώρες ε, δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια πλήρη μεταφορά. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μου αναλύουν τις πληροφορίες που έχουν στείλει τα κράτη-μέλη και δεν θα διστάσουμε να πραγματοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα βήματα και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε πλήρη μεταφορά και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις εξής εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρώτον, στι αρχές του 2016 θα υποβάλουμε την πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με βάση το άρθρο 20 της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη και η κοινωνία των πολιτών, όπως εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουν υποβάλει πληροφορίες στον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά της εμπορίας, όπως προβλέπει το άρθρο 20, και οι υπηρεσίες μου εκπονούν αυτή τη στιγμή τη σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή θα λάβει υπόψη και τη διάσταση του φύλου και συναφή ζητήματα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μία ενοποιημένη έκθεση για το άρθρο 23 της οδηγίας το 2016 επίσης. Η έκθεση αυτή θα αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη προκειμένου να τηρήσουν την οδηγία κατά της εμπορίας ανθρώπων. Επίσης θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των υπαρχουσών νομοθετικών διατάξεων που ποινικοποιούν το, την εμπορία και τους αυτούργους και μέτρα για την πρόληψη αποσόβηση τέτοιων εγκλημάτων και σχετικές προτάσεις. Η έκθεση αυτή επίσης θα λάβει υπόψη τη διάσταση φύλου της εμπορίας των ανθρώπων και θα συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ε, που αποτελεί το κίνητρο για τέτοιου είδους εκμετάλλευση. Η οδηγία πάταξης ε, της εμπορίας ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει νομικές υποχρεώσεις για τη μείωση της ζήτησης που αποτελεί το κίνητρο της εκμετάλλευσης. Και μάλιστα ε, σκοπεύει να ποινικοποιήσει και τους χρήστες των υπηρεσιών των θυμάτων. Η οδηγία για τις κυρώσεις των εργοδοτών ήδη ποινικοποιεί εκείνους που έσ χρησιμοποιούν θύματα εμπορίας υπηκόου τρίτων χωρών. Και μάλιστα οι υπηρεσίε μου έχουν αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για τη διάσταση φύλου στην εμπορία ανθρώπων σε ένα γνωστό ακαδημαϊκό Ινστιτούτο προκειμένου να, εξεταστούν, να εξεταστεί η διάσταση του φύλου στην εμπορία για ε, σεξουαλικούς σκοπούς και πρόταση μέτρων για να μειώσουμε τη ζήτηση που ενισχύει αυτή την εκμετάλλευση. Μάλιστα η μελέτη έλαβε επίση υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκφράστηκαν στο ψήφισμα του Φεβρουαρίου του, του 2014 για τα αποτελέσματα ε, της ε, πόρνειας ε, και την, τις συνέπειες τους στην ισότητα των φύλων. Η σχετική έκθεση θα ολοκληρωθεί φέτος, μέχρι τα τέλη του έτους. Και μάλιστα η στρατηγική μας θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016. Και όπως προβλέπετε στα ευρωπαϊκά θεματολόγια για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, θα υιοθετήσουμε μια στρατηγική και μετά το 2016. Και γι' αυτό θα έχουμε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους και σίγουρα θα κρατάμε συνεχώς ενήμερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να υποβληθεί μετά την προσέγγισή μας για την εποχή μετά το 2016. Κυρίες και κύριοι, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε έργο. Αυτό είναι σημαντικό και το οφείλουμε και στα θύματα αλλά και στην κοινωνία μας, στα παιδιά μας και στις επερχόμενες γενναίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρικά ιδιαίτερα που άκουσα ότι θα αναλάβετε συγκεκριμένα μέτρα για να δείτε ιδιαίτερα το θέμα του πόσο ευάλωτες είναι οι γυναίκες. Περνάμε τώρα στου ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η διακίνηση εμπορία ανθρώπων έχει γίνει πλέον η δουλεία της εποχής μας τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Το ΕΛΚ βεβαίως υποδέχεται θετικά το ότι θέλετε ακριβώς να δείτε τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Ανισχούμε όλοι, πρόκειται για σοβαρό οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακές διαστάσεις και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αντιμετώπιση με συνεργασία της αστυνομίας και της δικαιοσύνης μέσω της Europol, τη Eurojust και τη Frontex. Πρέπει να σπάσει αυτό ο κύκλο της ατιμορρησίας. Δεν πρέπει να μπορεί κανείς από αυτούς τους εγκληματίες να κρυφτεί πουθενά εντός και γύρω από την Ευρώπη. Ζητάμε λοιπόν να φέρετε γρήγορα την έκθεση για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση, γιατί όπως είπα, τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες που προκαλούν την εμπορία ανθρώπων, αλλά και βεβαίω η προστασία των θυμάτων κοριτσιών, γυναικών έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και βεβαίως πρέπει να μειωθεί και η ζήτηση. Πρέπει να καταστήσουμε υπεύθυνου και τους χρήστες. Η πλειοψηφία βεβαίω συνεχίζουν να είναι γυναίκες και παιδιά και όλο και περισσότερο μετανάστες. Οπότε η νέα σας στρατηγική, στρατηγική με κατά της ε, δραστηριότητας αυτής ε, πρέπει να έχει και την διάσταση του φύλου ποινικοποίηση και να παρακολουθείτε και τις χρηματικές ροές. Η ομάδα μας, κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσει να έχει μηδενική ανοχή κατά της εμπορίας ανθρώπων και βεβαίως θα έχει στην πρώτη γραμμή τα δικαιώματα του φύλου. Κανείς δεν θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης καθοδόν προς την ασφάλεια στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, κυρία Χάνιμπολ, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ βεβαίως καλωσορίζω τα όσα είπε ο κύριος Επίτροπος και την δράση που προανήγγειλε ότι δηλαδή σκοπεύεται να διασφαλίσετε ότι η ευθύνη θα αφορά και τους χρήστες και όχι τα θύματα των σεξουαλικών υπηρεσιών. Και όπως είπαμε όλοι πρόκειται κυρίως για ένα ζήτημα που πλήττει τις γυναίκες. Και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα πανευρωπαϊκά και να δούμε τις τακτικές ε, των διακινητών που φαίνεται πως ε, πάντα είναι ένα βήμα μπροστά στο ζήτημα αυτό της νέας δουλείας. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εγώ είμαι βουλευτής Λονδίνου που είναι ένας ε, προορισμός ε, για τους διακινητές και καθώς προετοιμαζόμαστε για το δημοψήφισμα για το αν θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ πως ε, το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων θα μας απασχολήσει. Ειδικά γυναίκες και παιδιά είναι ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και θεωρώ πως έχει ευρωπαϊκές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπιόρκ έχει τώρα το λόγο. Χάρηκα κύριε Επίτροπε που άκουσα ότι θα ζήτηση. Ποια είναι η ζήτηση όμως εδώ πέρα. Είναι βεβαίως και η προαγωγή και οι διοκτήτες οίκων αλλά και οι πελάτες. Και βεβαίως πρέπει να δούμε το ζήτημα της αγοράς. Και όπως είπε και η κυρία Χάνιμπολ, το σκανδιναβικό μοντέλο που ποινικοποιεί και την δραστηριότητα των προαγωγών αλλά και των πελατών έχει καταστήλει κατά πολύ την ζήτηση. Τι θα γίνει λοιπόν για να καταστήλουμε την ζήτηση για την αγορά γυναικών και κοριτσιών. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Διάβασα την έρευνα η οποία ανατέθηκε σε μια ομάδα λομπιστών οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα και ανισχώ ιδιαίτερα. Και δεν είναι σοβαρό και για να το πω και ομά δεν χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς και συνοριοφύλακες για αυτή τη δουλειά, χρειαζόμαστε λιγότερους οίκους ανοχής. Αναμένουμε λοιπόν έναν επικοδομητικό διάλογο για να γίνει, κάνουμε πραγματικά κάτι για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπούρς έχει το λόγο. Η ελευθερία μετακίνησης ε, μεταξύ των χωρών είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να ασκηθεί αυτή η εγκληματική δραστηριότητα. Τώρα αν τα θύματα είναι άντρες, γυναίκες, ε, κορίτσια ή αγόρια, το να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στα σύνορα προφανώς καθιστά πάρα πολύ εύκολη την ε, διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παραδέχεται πως αυτοί οι κανόνες βοηθάνε το οργανωμένο έγκλημα να διακινήσει όχι μόνο παράνομα αγαθά, αλλά και ανθρώπους. Όσον αφορά δε την έκθεση του 2015, λένε ξεκάθαρα πώς η ελεύθερη διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, από οργανωμένες ομάδες για να φέρουν μέσα ναρκωτικά, θύματα εμπορίας ανθρώπων, παράνομους μετανάστες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έκθεσή σας παραδέχεται πως η ελεύθερη μετακίνηση εντός των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης μειώνει τις πιθανότητες ανείχνευση. Η Eurostat λέει πως 68% των θυμάτων είναι γυναίκες. Πράγματι συγκλονιστικό όμως ο στόχος θα πρέπει να είναι να σταματήσει το φαινόμενο ε, ούτως ή άλλως, όχι να ανησυχούμε για την διάσταση του φύλου. Οι κανόνες λοιπόν της ελεύθερης μετακίνησης κάνουν την δουλειά των εγκληματιών πιο εύκολη. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάποια κάποιες προσπάθειες για να γίνει αδύνατη η δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων και οι τιμωρίες να είναι τέτοιες που να λειτουργούν αποτρεπτικά. Μόνο τότε θα σταματήσει αυτή η σύγχρονη μορφή δουλείας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπιτζότο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε για αυτό το σημαντικό θέμα, αλλά όχι ενώπιον 15 ανθρώπων. Είναι ταπεινωτικό. Όχι για μένα, αλλά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η διακίνηση των ανθρώπων είναι απαράδεκτη σε οποιαδήποτε μορφή της. Είναι τόσο, ε, υπάρχει τόση υποκρισία στην Ευρώπη. Ε, δεν μπορούμε να κρύψουμε την ε, κακή μας συνείδηση. Πρόκειται για ένα εμπόριο που αφορά την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα χθε έγκλημα. Το 2015 έφτασαν 250.000 ε, μετανάστες, οι οποίοι διέπλευσαν τη Μεσόγειο. 3.000 από αυτούς ε, πνίγηκαν ή χάθηκαν. Δεν θέλω, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η Αφρική και να είναι ε, γεμάτη από τις σημαίες του Ισλαμικού κράτους. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στις γυναίκες και στα παιδιά. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανθρωπιστικούς ε, διάβλους στις περιοχές σύραξης. Υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Έσαριτς. Τη δέχεστε? Ευχαριστώ. Συμφωνείτε ότι αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα είναι ε, κάτι το ε, σοκαριστικό και ίσως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι να υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος ε, ε, περνά τα σύνορα από την μία ή την άλλη πλευρά. Μπιτζότο. Σίγουρα θα πρέπει να ελέγξουμε τα σύνορα μας. Αυτό ζητούν οι πολίτες μας, αλλά δεν θα πρέπει να ε, φτάνουν, ε, δεν φτάνουν μόνο παράνομοι μετανάστες, φτάνουν και πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να τους ε, δεχτούμε όλους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τους ε, πρόσφυγες, αλλά θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να ζήσουν στην Αφρική και όχι να μεταβαίνουν στην Ευρώπη. Στο κατάλογο ομιλητών, κυρία. Είχατε ήδη την ευκαιρία να μιλήσετε, δεν μπορώ να σας δώσω δυνατότητα να υποβάλλετε ερώτηση. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή τον κύριο Φουντούλη. Δεν χωρά καμία αμφιβολία πως η εμπορία ανθρώπων είναι ένα φαινόμενο κατάπτυστο και απεχθές, μία βόμβα στα θεμέλια του αξιακού συστήματος της Ευρώπης. Αδιαπραγμάτευτη στάση μας θα πρέπει να είναι η συνεχής προσπάθεια όχι για τον περιορισμό του φαινομένου αλλά για την πλήρη εξάλληψή του. γεγονό είναι πω στη σύγχρονη εποχή οι γυναίκε είναι εκείνε που πλήττονται περισσότερο από αυτέ τι πρακτικέ για λόγου που όλοι γνωρίζουμε. δυστυχώ έχουν έρθει στο φω πάρα πολλέ υποθέσει στι οποίε υπήρξε σιωπηρή ανοχή ή ακόμα και συνενοχή κρατικών λειτουργών. πρέπει να υπάρξει εκ μέρου μα μια αποφασιστική δράση για την πάταξη των κυκλωμάτων που επωφελούνται από την εμπορία ανθρώπων. δεν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ακόμα ηθικολογικό κείμενο όμορφο στα λόγια αλλά με κανένα πραγματικό αντίκρισμα. πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε μέσο πίεση προ τα κράτη μέλη ώστε να μην υπάρξει καμία ανοχή στου διακινητέ. όταν κάποιο προσβάλλει με τέτοιο βάναυσο τρόπο τι αξίε και τι αρχέ των ευρωπαϊκών λαών πρέπει να έρχεται αντιμέτωπο με τι αυστηρότερε δυνατέ ποινέ. η ένωση οφείλει να δεσμευτεί στου λαού τη πω θα τσακίσει τη διεθνή αυτή μαφία θα γκρεμίσει τα εμπόδια μέχρι να επιτευχθεί η πλήρη εξάλληψη του δικτύου είτε αφορά εμπορία γυναικών είτε αφορά εμπορία και εκμετάλλευση οποιαδήποτε ανθρώπου. σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χέντ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η οδηγία για την εμπορία ανθρώπων του 2011 αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα ε, συγκεκριμένο ε, σεξοκεντρικό έγκλημα. Αυτό που αφορά την εμπορία ανθρώπων αφορά ε, ένα έγκλημα που πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια, τα μικρά κορίτσια ή τις εφήβους που αγοράζονται στην ουσία από τους άνδρες. Δεν πρέπει να δεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις της έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά στα κράτη-μέλη η οδηγία του 2011. Και αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να απαιτήσει κανείς. Πιστεύω ότι η παράνομη ε, διακίνηση των ανθρώπων είναι κάτι το αποτρόπαιο. Θα πρέπει πλέον να δράσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζουμπέρ είναι η επόμενη αμελήτρια. Είναι κατεπήγον και απαραίτητο καταρχήν να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία για την εμπορία των ανθρώπων. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, που είναι αυτά της Eurostat, αναφέρονται στο 2012. Ε, ενώ είχαμε ε, ε, δεινές καταστάσεις οικονομικές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδείνωση της κατάστασης της πολιτικής σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Με όλες αυτές τις επιδεινώσεις η σημερινή πραγματικότητα είναι ακόμη πιο απάνθρωπη και σκληρή. Το 2012 74% των θυμάτων ήταν γυναίκες και 13% του συνόλου ήταν κορίτσια. 66% των ανθρώπων που ήταν θύματα εμπορίας έγινε και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 96% αυτών ήταν γυναίκες. Όπως αναγνωρίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων και της ε, πορνείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης υπάρχει άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της πορνείας και της ε, εμπορίας γυναικών. Ένα μεγάλο τμήμα της εμπορίας αυτές θα πρέπει να, να καταργηθεί και φυσικά να ποινικοποιήσουμε όσους ε, ζουν βιοπορίζονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Αυτό. Κύριε Πίτροπο, σήμερα στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε τις πιο σοβαρές ε, περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων που πλήττουν δυστυχώς τις γυναίκες. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλες τραγωδίες που χρησιμοποίησε και ο τύπος. Υπάρχουν πολυπληθείς ε, περιπτώσεις. Πολλές είναι οι γυναίκες οι οποίες στην ουσία μπαίνουν στα πλοία ε, σε κατάσταση εγκυμοσύνης για να μπορέσουν να γεννήσουν στην Ιταλία ή σε μια άλλη χώρα. Η Europol μιλά για 30.000 διακινητές που βρίσκονται πίσω από τη μετανάστευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε για παράνομη δραστηριότητα και κέρδη που υπερβαίνουν ε, τα κέρδη από την πώληση όπλων. Είναι η καλύτερη business δηλαδή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη σύγχρονη τραγωδία διακίνησης ανθρώπων. Η κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Oh, Επιτρέψτε μου Sorry. Ε, ε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έκανα εγώ λάθος. Το λόγο έχει η κυρία Φορέντσα. Κυρία Φορέντσα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το αίτημα προς την Επιτροπή, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ε, ελέγξουν τη σωστή εφαρμογή του δικαίου και το μηχανισμό αυτό να υποπτεύσει η Επιτροπή. Θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά, διότι θα πρέπει το δικαίωμα της ε, ε, μη διακίνησης των, ε, των γυναικών και το δικαίωμα να ορίζουν τη ζωή τους όπως θέλουν είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει να υπάρχει και σωστή εκπαίδευση και άπτεται του ζήτηματος. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, τρομοκρατούμε τις γυναίκες θα πρέπει να έχουν μια πολύ σωστή προσέγγιση ως προς τον ίδιο τον εαυτό τους, το σώμα τους. Ένα 70% των θυμάτων είναι γυναίκες, αλλά αυτοί που ε, εκμεταλλεύονται τις γυναίκες είναι άνδρες και δεν θα πρέπει να δούμε τις γυναίκες σαν απλά σώματα. Είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι με ψυχή. Ε, ευχαριστούμε πολύ. κυρία συμφωνώ μαζί σα, και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λόγω τη κατάσταση επιτρέψτε μου να είμαι κατηστή. Το θέμα τη σημερινή συζήτηση μου είναι ευωτήτατα λιβαρό. Θα μοιραστώ ένα δικό μου στοιχείο στην έκθεση που ετοιμάζω για λογαριασμό τη Επιτροπή ΦΑΜ για το οικιακό προσωπικό και εργαζομένε φροντίδες διαπίστωσα με τλίψη πώ ένα κομμάτι αυτού του τομέα εργασία τροφοδοτείται από την παράνομη εμπορία και διακίνηση ανθρώπων. Ανθρώπινες ψυχές που χωρίς να ξέρουν συνένεσαν στο να γίνουν ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα του τράφικινγκ, ακολουθώντα διακινητέ που του υπόσχονται καλέ δουλειέ. Ψυχέ που καταλήξαν θύματα σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση. Και η Επιτροπή τι κάνει για να προστατεύσει τα θύματα αυτά, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκε. Βρίσκεται για άλλη μια φορά πίσω από εξελίξει, καθυστερώντα ακόμα και τα και να αξιολογήσει τα μέτρα που ήδη ζήτησε από τα κράτη μέλη να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης ανθρώπινων ψυχών. φυσικά και τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη γι' αυτό γιατί επιτρέπουν στην πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης να είναι αντιφατική και ορισμένε φορέ υποκριτική στο θέμα του τράφικινγκ. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φαίνεται αυστηρή σε ό,τι αφορά το τα παράνομη διακίνηση, ταυτόχρονα με τα μεταναστευτική τη πολιτική, όμω όπω αυτή εφαρμόζεται σήμερα, αμέσω επιτρέπει το φαινόμενο. Κλείνοντα, τι νόμιμε οντού μετανάστευση σπρώχνουν την συναγκαλιά παράνομων διακινητών χιλιάδε γυναίκε. Λυπάμαι που το διαπιστώνω, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει στην άντιση του φαινόμενου του τράφικινγκ. Έχει όμω μια ευκαιρία να ανακόψει το φαινόμενο πριν να είναι πια πολύ αργά. Πώ αν αξιολογήσει και να θεωρήσει άμεσα τα μέτρα εκείνα που θα τη επιτρέψουν να επιτύχει του στόχου που έθεσε στη 2012-2014. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμω, χωρί συνοχή μεταξύ της μεταναστικής πολιτική της πολιτικής για το τράφικινγκ, της αναλύσης της φιλελευθερικής διαστάσης το φαινόμενο να βρεθούμε άλλη μια φορά μάρτυρες περιστατικών επιστεύτης φρίκης με πολιτισμένη Διακόπτη την κυρία Κούνεβα η, ομιλή, η πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε την συζήτηση με γεγραμμένους ομιλητές. Θα περάσουμε στο Catch the Eye. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους ε, όσοι τον ζήτησαν, αλλά θα είμαι πολύ αυστηρή στην τήρηση του χρόνου και θα σας διακόπτω με το που θα ξεπερνάτε το λεπτό. Η κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ τον Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δράσεις και τις προσπάθειές τους για την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων. Η οδηγία για το τράφικινγκ απαιτεί καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Ε, θα θέλαμε κατεπηγόντως να προστατεύσουμε παρκώς και τα θύματα και να ε, αναζητούμε τους αυτούργους, γιατί δεν ε, ποινικοποιούμε τα θύματα, αλλά τους μαστροπούς και τους διακινητές. Επίση, υπάρχουν διακινητέ που επεκτείνουν τι δραστηριότητέ του χρησιμοποιώντα το διαδίκτυο. Θα πρέπει επίση να δούμε και να ενισχύσουμε τι ε, διοικητικέ δομέ με τι οποίε έρχονται σε επαφέ ε, τα θύματα του τράφικινγκ για να μπορούν να καταγγέλλονται τέτοιε περιπτώσει ε, και επίση να δούμε και επιχειρήσει που εποφελούνται από θύματα. Σα ευχαριστώ. Κυρία Μίλτση, έχει το it-traffikar tan-nies hi problema gravi u Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα πολύ ενισχυτικό πρόβλημα. Χιλιάδες άνθρωποι πολλούνται στην ε, Ευρώπη και δουλεύουν με τρόπο αναξιοπρεπή. Και βεβαίως ε, όλα αυτά ενισχύουν το οργανωμένο έγκλημα και το πρόβλημα συνεχώς ε, διωγγώνεται. Τη στιγμή που μιλάμε, γυναικόπαιδα πραγματικά χάνουν την ε, ζωή τους με τρόπο τραγικό. Πρόκειται για μια σύγχρονη μορφή δουλείας, σκλαβιάς και παραβιάζει κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Γι' αυτό τον λόγο και άλλους απευθύνω έκκληση στην ε, Κομισιόν ε, και στα κράτη-μέλη να είναι άτεγκτοι και να λάβουν υπόψη την διάσταση του φύλου. Τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και κοριτσιά. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εμπορία και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι έγκλημα και ως τέτοιο πρέπει να τιμωρείται. Έχει αποκτήσει μια σημαντική διάσταση τώρα εν ώψη των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το ζήτημα των δουλεμπορικών κυκλωμάτων τα οποία υπάρχουν κυρίως στην Τουρκία όπου δρούν. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από την Συρία να έχουν μεταφερθεί στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά έτσι μόνοι τους. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το καλοκαίρι πήγα στο Κουσάνταση γιατί ήθελα πραγματικά να δω τι γίνεται ενώ απέναντι στη σάμο υπήρχαν χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην πλευρά της τουρκίας δεν υπήρχε ούτε ένας διότι γίνεται πολύ οργανωμένη η διακίνηση διότι τους εφοδιάζουν με σωσίβια και βάρκες διότι τους έχουν σε οργανωμένες κατασκηνώσεις. πρέπει να γίνει μια αποστολή μια fact finding mission για να δούμε το ζήτημα της δουλεμπορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο, κύριο Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπορία ανθρώπων, το τράφικινγκ, ε, είναι σήμερα σίγουρα μια από τις πιο κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γινόμαστε μάρτυρες αυτής της ε, καταπάγεδων καθημερινά. Το τράφικινγκ, ε, η εμπορία των ανθρώπων, μαστίζει κυρίως τις γυναίκες. Αυτές είναι τα πιο ευάλωτα θύματα του τράφικινγκ. Και αυτό δείχνει ε, τι υποκρισία υπάρχει και τι κακοβουλία ε, από όσους, ε, όλους εκείνους που ανέχονται αυτή την κατάσταση. Πριν από λίγο μιλήσαμε για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και τώρα μιλούμε για την καταπάτηση αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με την εμπορία. Και παρόλο που υπάρχει, υπάρχουν σχετικές ε, διατάξεις, δυστυχώς πολλές ε, χώρες μέλη ακόμη δεν τις έχουν εφαρμόσει. Κρίμα. Θα πρέπει να μιμηθούμε το σκανδιναβικό μοντέλο ε, λύση των προβλημάτων, γιατί έχει αποδείξει και εμπράκτος ε, τα πλεονεκτήματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συζητάμε ένα πανάρχαιο πρόβλημα. Την δουλεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση σε έναν κόσμο όπου απεγνωσμένοι άνθρωποι μεταναστεύουν σε τεράστιους αριθμούς. Το περιβάλλον είναι τέλειο για τους διακινητές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Χρειάζονται αυστηρή έλεγχη στα σύνορα, βαριές τιμωρίες για τους διακινητές ανθρώπων, συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων κρατών μελών για να αντιπαλέψουμε αυτό το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δικαίου και συγκεκριμένα του διεθνούς δικαίου προωθείται καλύτερα με αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους. Έχουν υποχρέωση απέναντι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά που διακινούνται με αυτόν τον άσχημο τρόπο να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Πρότσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Οπωσδήποτε συμφωνώ πως η συμπεριφορά αυτή είναι καταδικαστέα. Είτε μιλάμε για διακίνηση γυναικών, είτε για πορνεία, ε, την εκμετάλλευση στο διαδίκτυο, όλα αυτά είναι αποκουστικά. Από την άλλη, ε, κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στους μετανάστες και σήμερα το πρωί εξεπλάγιν όταν είδα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην έκθεση Κέλλερ και οι συνάδελφοι που θέλαν ε, και στήριξη και γυναίκες από την ομάδα μου δεν στήριξαν αυτή την έκθεση και μετά μιλάνε για υποκρισία. Μα πώς ζητάτε ε, ευρωπαϊκή ελεγγύη και μετά κάποιες και γυναίκες μάλιστα δεν έκαναν ε, τα απαραίτητα για να βοηθήσουν οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας. Είναι πραγματικά καταδικαστικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε πλήρη στοιχεία για τη διακίνηση ανθρώπων. Και όπως είπε και η συγγήτρια, τα στοιχεία είναι πολύ ψηλότερα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας γιατί τα θύματα φοβούνται να μιλήσουν και εδώ θα πρέπει να δράσουμε κύριε Επίτροπε να δούμε όχι μόνο την εποπτεία, αλλά να βρούμε και λύσεις για να προστατεύσουμε τα θέματα. Χρειάζεται απαιτητική εποπτεία, αλλά δεν επαρκεί εάν δεν βρούμε λύσεις και φτάσουμε στη ρίζα του κακού. Θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις και καταδίκη αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να καταδικάσουμε τους ε, ε, διακινητές. Μιλάμε για μια σύγχρονη, σύγχρονη δουλεία. Θα πρέπει να μας πείτε ποιες είναι οι δύο χώρες που δεν, ε, έκαναν, δεν έλαβαν τα σωστά μέτρα. Σκρίπεκ. Κύριε Σκρίπεκ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οπωσδήποτε η πορεία ανθρώπων είναι παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να δούμε και τις νέες μορφές ε, ε, πορεία ανθρώπων μεταξύ των ε, οποίων και την ε, λεγόμενη ενοικίαση μήτρας. Στην αρχή μιλούσαμε μόνο για εμπόριο αρίων, αλλά τώρα πλέον βλέπουμε πως ε, ε, κάποιες γυναίκες μένουν έγκυος για λογαριασμό άλλων. Βλέπουμε επίσης πως πρέπει να ερευνηθούν οι δραστηριότητες του IPPF ε, της International Plant Parenthood Federation. Μέχρι τότε είμαι κατά οποιασδήποτε χρηματοδότησης αυτής της οργάνωσης. Δεν επιτρέπεται να κλείνουμε τα μάτια. Δεν είναι δυνατό να πραβιάζεται έτσι το δίκαιο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε κυρία Πόστ. Thank και κύριοι. Α, όχι, ο κύριο Φρουνζουλίκα Η κυρία Πόστα έχει το λόγο και μετά εσείς ε, κύριε Φρονζολικά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διακίνησης και να δούμε κατά πόσο αυτοί που αγοράζουν τις υπηρεσίες ε, ε, δεν θα πρέπει να διωχθούν. Πρόκειται για μία αλληλένδετη πορεία δραστηριοτήτων θα πρέπει να δούμε ποιος ε, χρησιμοποιεί αυτές τις ε, δυνατότητες. Νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην εφαρμογή του, της οδηγίας από τα κράτη-μέλη. Επίσης, σε περίπτωση συνεχόμενου βιασμού, κατά συρροή βιασμών, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα νέα αυτά θύματα δεν έχουν το κουράγιο να καταγγείλουν. Σε αυτή την περίπτωση όμως, αν γίνει η καταγγελία, θα πρέπει τουλάχιστον να μπορούν να, έχουν, να πάρουν άδεια παραμονής. Ο με συγχωρείτε, δεν άκουσα καλά. Σας ευχαριστώ. Η εμπορία ανθρώπων, κύριε και κύριοι, είναι σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος που πρέπει να καταπολεμήσουμε με κάθε μέσο. Γυναίκες, άντρες και παιδιά διακινήθηκαν με διάφορους τρόπους και απαιτούν την στήριξή μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια σαφή διάσταση του φίλου και να δέσουμε προτεραιότητα στα θύματα και τις ανάγκες τους. Η προτεραιότητά μας που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να επικεντρωθεί στα θύματα και να αποθαρρύνει την ζήτηση για κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βεβαίως και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, πως η πρόταση αυτή έχει στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των διαφόρων εμπλεκομένων. Οπότε τα κράτη-μέλη πρέπει να σεβαστούν τις προθεσμίες μεταφοράς και συμμόρφωσης και η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία και Δεν Τελειώσαμε συγχωρείτε με τη διαδικασία και HDI. Τον λόγο έχει ο κύριος Αβραμόπουλος. Κύριε Επιτροπέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με κάτι πιο γενικό. Βλέπω πως κάποιοι βουλευτές χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να επιτεθούν σε ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την ελευθερία μετακίνηση σε μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα. Θα επαναλάβω πως η Σέγγεν είναι τμήμα της λύσης, όχι του προβλήματος. Με το να εκμεταλλευτούμε πλήρως τους κανόνες της Σέγγεν, ε, μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τα σύνορά μας. Τώρα, στο θέμα μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για αυτή την σύντομη αλλά ουσιαστική συζήτηση. Προφανώς συμφωνούμε. Η διάσταση του φίλου πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Να είμαι σαφής. Η εμπορία ανθρώπων είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά θύματα της εμπορίας ανθρώπων ακόμα και αυτό είναι απαράδεκτο. Κυρία Μπιέρκ, όπως πολύ καλά ξέρετε, η ποινικοποίηση της ζήτησης των χρηστών που εν γνώση τους χρησιμοποιούν θύματα εμπορίας θεωρείται ένα μέτρο μείωσης της ε, ζήτησης. Η οδηγία δε παροτρύνει τα κράτη-μέλη να σκεφτούν κάποια μέτρα ε, όταν γνωρίζουν πως ένα άτομο είναι θύμα τράφικινγκ. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν την ε, χρήση και τους ε, χρήστες ε, ατόμων που γνωρίζουν ότι πρόκειται για θύματα εμπορίας. Απλά λέει ότι θα πρέπει να το εξετάσουν. Και κάποια από αυτά το κάνουν βεβαίω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε αναζητούμε τρόπους να μειώσουμε την ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει δράση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν το τι έχουμε κάνει καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της στρατηγικής κατά της εμπορίας ανθρώπων και βεβαίως σκοπεύω να ανταλλάξω μαζί σας απόψεις για τη νέα στρατηγική πριν την υιοθέτησή της του χρόνου. Σας ευχαριστώ. La discussione è chiusa.